έλαβα από την Επιτροπή ΦΑΜ ένα αίτημα διαβούλευση με την ε, ΟΚΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για την προετοιμασία μιας έκθεσης πρωτοβουλία για την κατάσταση και τα δικαιώματα των γυναικών με ε, αναπηρίε. Αν εντό 24 ώρων καμία πολιτική ομάδα ή αριθμός ε, βουλευτών ε, ίσως με το κατώτατο όριο δεν ε, φέρουν αντιρρήσεις θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία διαφορετικά θα γίνει η ψηφοφορία και θα ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια ότι την ε, Τετάρτη